Εδώ προδίδεται το Κοινοβούλιο γιατί χειροκροτείται πραγματικά ε, και επιθυμείται για το κλιματικό κατεπήγον, ενώ στην πραγματικότητα πρημοδοτείται τι ε, πολυεθνικέ που ρηπαίνουν τη φύση. Είναι λοιπόν ανάγκη να δούμε και να αντιμετωπίσουμε κατάπατσα την κλιματική καταστροφή, να ξεκινήσουμε απαντώντας, αφήνοντας το φυσικό αέριο στη γη εκεί που ανήκει. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μόντι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ καταψήφισα τον κατάλογο αυτόν διότι υπάρχουν πάρα πολύ, πολλά έργα που περιλαμβάνουν ορυκτά καύσιμα. Ακόμη και αν επρόκειτο για μια μεταβατική περίοδο, ε, ε, πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτά τα έργα άπαξ και οικοδομηθούν και ολοκληρωθούν έχουν ένα κύκλο ζωής 40-50 ετών. Δεν μπορούμε μετά το 2050 να έχουμε ακόμα ορυκτά καύσιμα στο ενεργειακό μας ε, μείγμα. Ε, έρχεται σε αντίθεση με τις διακηρύξεις μας. Σε περίπτωση που τεθούν σε περαιτέρω επεξεργασία αυτά τα έργα, θα ήθελα η Κομισιόν να λάβει υπόψη της αυτό που έχει πει το Κοινοβούλιο για την κλιματική έκτακτη ανάγκη που έχουμε διακηρύξει. Έχουμε Πολάκης και επανειλημμένος ε, τονίσει ότι εμείς υποστηρίζουμε τη Συμφωνία των Παρισίων και μια ουδέτερη από άποψη άνθρακα ε, Ευρώπη το 2050. Ο κύριος Ρόντζα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Η ψηφοφορία αυτή πραγματικά ήταν μια εξαιρετική είδηση για πολλά κράτη-μέλη, διότι το φυσικό αέριο είναι ένα αγαθό αναγκαίο και είναι και μια βιώσιμη πηγή ενέργειας για πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων πολλών μετακομμουνιστικών χωρών. Εμείς, ε, ναι, επενδύουμε στο φυσικό αέριο και αυτό βοηθά εμάς, τις μετακομμουνιστικές χώρες, να εγκαταλείψουμε το παλιό ρηπογόνο ενεργειακό μα σύστημα. Και χάρη σε αυτήν την ψηφοφορία, σε αυτό το ψήφισμα, το Κοινοβούλιο κατέδειξε ότι μπορούμε να βρούμε συμφωνία ε, ανάλογα με, το, με την αφετηρία του καθενός και του στόχου του. Έτσι θα μπορέσουν λοιπόν να χρηματοδοτηθούν ε, αγωγή ε, φυσικού αερίου από την Ορβηγία, τις Βαλτικές χώρες, την Πολωνία, την Τσεχία, τη την Σλοβακία. Πρόκειται για συστήματα φυσικού αερίου που θα χρησιμοποιούν υγροποιημένο φυσικό αέριο και θα μας βοηθήσουν στην απόκτηση της ε, ανεξαρτησίας μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σίντσης έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Υπάρχει ένας ολόκληρος κατάλογος από έργα κοινού ενδιαφέροντος και ε, ο σταθμός στο Κίρκ. Θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά πριν ε, τα υλοποιήσουμε όλα αυτά και εάν βρεθεί κανείς σε ατυχή θέση όπως η Κροατία, αυτά τα μεγάλα έργα μπορεί πραγματικά να καταστρέψουν το περιβάλλον ε, και τις δικές μας ειδικές γνώσεις με την χρήση της τεχνολογίας. Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να είναι επιζήμια και υπάρχουν πολλά έργα που απειλούν τις τοπικές οικονομίες ε, σε χώρες όπως η Κροατία και Ήδη πληρώνουμε πολλά για τη διαχείριση των αποβλήτων, για το νερό και την υδροδότηση. Η Κροατία είναι μια χώρα απομακρυσμένη στην Ευρώπη. Έχουμε πολύ ακριβή ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να περάσει από την Αυστρία η παραγωγή της από άλλε χώρε. Πληρώνουμε ήδη πάρα πολλά για τα έργα ηλεκτροδότησης. και αυτό που έχω να πω είναι όχι ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο κύριος Βασική εσωτερική και μεταρρυθμιστέ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κατεψήφισα αυτήν την αντίρρηση. Γιατί θα πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτήν την παραλογή πολιτική. ψηφίζετε κατά του άνθρακα, ψηφίζετε κατά του φυσικού αερίου, αλλά κάνετε υπεργολαβία την απασχόληση και εκτός Ευρώπης. Καταψηφίζετε τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και την ευημερία των Ευρωπαίων. Κυρίως από όλα αυτά θίγονται οι χώρες Ανατολικής Ευρώπης. Μια χαρά είναι η καθαρή ενέργεια. Ωραία όλα αυτά τα όνειρα, αλλά, αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου όπως τα λέτε και δεν λάμπει ο ήλιος τη νύχτα. Λέγονται πάρα πολλά πράγματα που δεν στέγουν οι, οι οικολόγοι. Κούμπουλα Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτός ο κατάλογος των κοινών ε, έργων ή των έργων κοινών ενδιαφέροντος ε, έχει σχέση με ένα ευρύτερο θέμα, με έναν κανονισμό που μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέλει να τον αναθεωρήσει προς το καλύτερο ε, τα δίκτυα, ιδίως τους μηχανισμούς διασύνδεσης. Εν προκειμένου υπάρχουν κάποια κριτήρια που θα βοηθήσουν την καταπολέμηση αλλαγής του κλίματος, οπότε το μήνυμά μας ε, με την ψήφα μας είναι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θέλουμε αυτή η λίστα να αντιστοιχεί με τους στόχους μας και έτσι να έχουμε μια οικονομία χωρίς ε, χρήση άνθρακα. Δεν είναι τέλειος αυτός ο κατάλογος, αλλά τον ψήφισα. Τα τρία τέταρτα αυτών των έργων θα βελτιώσουν το ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτό είναι σημαντικό και άρα θα πρέπει αυτό να έχουμε υπόψη μας. Δεν ξέρω αν ακόμα έχουμε κάποια έργα που δεν έχουν πάρει την χρηματοδότηση όπως θα τα κράτη-μέλη. Αλλά νομίζω ότι τώρα θα βελτιωθούν τα πράγματα. Ευχαριστούμε για το έλκο κύριος Κέλλη είναι ένα από τους 430 ε, ε, ε, βουλευτέ που ψήφισαν αυτή την αντίρρηση για την λίστα και το πιστεύω ότι αυτά τα έργα είναι πάρα πολύ σημαντικά, ούτω ώστε να έχουμε μια εύρυθμη ενεργειακή αγορά και θεωρώ ότι έτσι θα έχουμε καλύτερη προμήθεια και προσφορά ενέργειας, απασχόληση και ανάπτυξη στις περιοχές που καλύπτονται όλα αυτά που μια δέσμη και έχουμε εδώ ένα σωρό σημαντικά πράγματα για τους Ευρωπαίους, σημαντικά έργα και έτσι θα προχωρήσουμε προς την Ελληνική Ένωση και στην Ιρλανδία έχουμε τέτοια όπως ε, τον κελτικό σύνδεσμο και επίσης ε, και έργα εξηλεκτρισμού, σύνδεση με το Ηνωμένο Βασίλειο και διάφορους ηλεκτρικούς σταθμούς ε, οπότε προχωρούμε προς τον στόχο μας να έχουμε 70% ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2030. Έχουμε τώρα και κάποια έργα για το φυσικό αέριο που είναι σημαντικό στην ε, κλιματική αλλαγή, στην ενεργειακή αλλαγή και να δούμε τι θα γίνει με τις μεταφορές και άλλους ε, τομείς όταν αντικαταστήσουμε τα ορυκτά κάψιμα και τον άνθρακα. Η Οπότε τελείωσε αυτή η ενότητα αγοριτών και πάμε στο επόμενο θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό που είναι η στρατηγική της Ένωσης για τον τερματισμό της πρακτικής ακροτηριασμού των ε, γεννητικών οργάνων των γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρακαλώ. Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα αυτό και μίλησα για αυτό το θέμα το 2011 όταν η Ιρλανδία πρότεινε ε, νομοσχέδιο στο Κοινοβούλιο για την απαγόρευση αυτής της βάρβαρης πρακτικής στη χώρα. Ανεξάρτητα από θρησκευτικές πεπιθήσεις του καθενός, αυτό έρχεται σε αντίθεση με το θεμελιώδη δικαίωμα της σωματικής ακαιρεότητας και της υγείας. Από αυτή την άποψη λοιπόν χαιρετίζω αυτό το ψήφισμα και καλώ την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να προστατεύουν τους ανθρώπους τους σε όλη την επικράτεια της Ένωσης, να έχουν εύρωστη νομοθεσία μέσω των εθνικών τους κοινοβουλίων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν σημαντικότατες ε, κυρώσεις εναντίον των ανθρώπων εκείνων που συμμετέχουν ή επιδίδονται σε αυτή την πρακτική. Και θα πρέπει ταυτόχρονα να έχουμε υπηρεσίες υποστήριξης και υγειονομικής περίθαλψης ώστε τα, τα θύματα του ακροτηριασμού να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν υποστήριξη και βοήθεια εφόσον τη χρειάζονται, λόγω της ε, βλάβης που έχει προκληθεί στην ε, υγεία τους. Και καλό και τα Εθνικά Κοινοβούλια να θεσπίσουν σχετική νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαριανή για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποψήφισα το ψήφισμα αυτό, διότι η κλειτοριδεκτομή είναι μια βία πράξη που πολλές φορές έχει να κάνει με την εσφαλμένη και στρεβλωμένη αντίληψη σε πολλές Ισλαμικές κοινότητες. Εδώ λοιπόν αυτές οι πρακτικές που έχουν εξαχθεί ε, στο ευρωπαϊκό εδαφός ε, έχουν να κάνουν με τη μαζική μετανάστευση και πραγματικά έχουν σοκάρει τις κοινωνίες μας. Διαφορετικές ε, κουλτούρες με διαφορετικά ήθη και έθιμα είναι πραγματικά δείγμα αφέλειας από μας. Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχτεί τέτοιες προκατάσεις προκαταλήψει, ιδεολογίες, ε, που οι προκαταλήψεις που αναφέρονται στο ψήφισμα. Θα πρέπει να ζητήσουμε την κατάργηση αυτών των πρακτικών που πραγματικά ε, ε, εκτραχυλίνουν την ανθρώπινη φύση. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε για τον ε, οικουμενικό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι να τα επιτρέπουμε αυτά στην επιρρό μα. Είναι χιλιάδε οι γυναίκε που απειλούνται από αυτή την πρακτική στην επιρρό μα, μια πρακτική που τώρα την αγνοούσαμε, για να εφαρμόσουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική ε, προάσπιση των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων και του ευρωπαϊκού τρόπου ζωή. Αυτό θα πρέπει να προαχθεί, γιατί θα πρέπει να χτυπήσουμε χτυπήσουμε τα αίτια. Τα αίτια είναι βεβαίω η έλλειψη ελέγχου των ε, πηγών τη μετανάστευση και ο ε, πολιτιστικό μεσαίωνα, τον οποίο θα, θα επιστρέψουμε εάν ε, αυτέ οι ασφαλμένε πρακτικέ συνεχιστούν. Για το, ε, υπερψήφισα το ε, ψήφισμα αυτό. Ευχαριστούμε και πάλι από την, κυρία, από την ID, κυρία Ζωρό, αλλά δεν την βλέπω στην αίθουσα, οπότε περνάμε στην επόμενη ομιλήτρια, την κυρία Πελτιέ από την και αν η κυρία Ζωρόν επιστρέψει θα πάρει το λόγο μετά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ χαίρομαι που εγκρίθηκε το ψήφισμα αυτό. Υπερψήφισα προφανώς ε, διότι μετά την έγκριση του ψηφίσματος για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ε, τον Νέα του 2019 νομίζω ότι πρέπει να υποστήλουμε αυτό το ε, χειρό μήνυμα σε ό,τι αφορά τις βίες πράξεις κατά των γυναικών και τις ισότητα ανδρών γυναικών. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε συμπεριλάβει μεταξύ των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης την εξάλληψη των μορφών μορφών ε, γενετικής βίας ως το 2030 βλέπουμε ακόμη ότι η κλειτοριδεκτομή αφορά 6 ε, εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίω και 200.000 200 ε, εκατομμύρια γυναίκες στον κόσμο και χιλιάδες στην Ευρώπη. Εδώ λοιπόν η κλειτοριδεκτόμη είναι πραγματικά επίθεση στο γυναικείο σώμα και πνεύμα. θα πρέπει μακροπηρεασμός των γυναικείων ε, γενετικών οργάνων να ε, γίνει αποδεκτό ως ε, φαινόμενο έλλειψη ισότητα ανδρών και γυναικών και δεν μπορούμε, όπω και ο κύριο Μαριανή, να το συνδέουμε μόνο με τη θρησκεία. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε την πρόληψη και την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών κατά πρώτον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Πελτιέ. Και η κυρία Βυσνιεύσκα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε συνάδελφοι, είμαι τελείως αντίθετη σε κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών, ιδίως ε, τον ακροτηριασμό των γυναικείων γενετικών οργάνων. Είναι μια πρακτική που τη βλέπουμε να εφαρμόζεται σε κάποια ευρωπαϊκά κράτη. Είναι μια μορφή κτηνώδης να υποβαθμίζονται οι γυναίκες. Πληγώνουμε το ίδιο του το σώμα. Γι' αυτό το λόγο καταψήφισα ε, μάλλον καταψήφισα το ψήφισμα αυτό και επειδή ε, κάποιες πολιτικές ομάδες θα να περάσουν τη δική του πρόπτικη, ορισμένες τροπολογίες δεν τι ψήφισα. Η κλειτοριδεκτομή είναι κάτι που θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, κρυζωθεί. Ε, θα πρέπει να υπάρξει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των ε, παιδιών και των νέων. Και να κοιτάξουμε τι εκφράσει που χρησιμοποιούμε σε σχέση με την αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία. Εδώ μιλάμε για τον ακροτεριασμό των γυναικείων οργάνων και τη φροντίδα που χρειάζονται αυτέ οι γυναίκε κατόπιν ω ασθενεί. Ε, θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε τι εκφράσει έχουν χρησιμοποιηθεί στο ψήφισμα κατά των αμβλώσεων. Δεν συμφωνώ με το σημείο 20, όπου μιλάμε για την κύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Ευχαριστούμε, κυρία Άντερσον. Επόμενη. Ευχαριστώ. Το ψήφισμα αυτό έχει ως ε, στόχο την καταπολέμηση του ε, ακροτηρισμού των ε, γυναικείων γεννητικών οργάνων. Δυστυχώς όμως για άλλη μια φορά μιλάμε για ένα αδιανό πουκάμισο. Διότι την, τον ακροτηριασμό δεν μπορείς να τον καταπολεμήσεις εκφωνώντας λόγους ή βάζοντας αυτοκόλλητα στο πέτο του κανείς. Αντίθετα, εγώ είχα είχα αποτύχει με μια πρωτοβουλία μου, η οποία είχε ως στόχο να διευρύνουμε την ε, Σύμβαση Κωνσταντινούπολης. Ούτε θα βοηθούσε το να δώσουμε προτεραιότητα όσον αφορά την υποβολή αίτησης ασύλου ε, ε, σε κορίτσια που έχουν υποβληθεί σε αυτή την απανθρώπη, απάνθρωπη μάλλον πρακτική. Γιατί στην ουσία αυτό θα είναι σαν ένα διαβατήριο, σαν ένα κίνητρο να γίνεται ακροτερισμός ώστε να στέλνονται μετά τα παιδιά. Αυτό δεν γίνεται. Γνωρίζουμε όλοι ότι το Ισλάμ είναι μια κουλτούρα η οποία περιφρονεί τις γυναίκες. Όποιος δεν το λέει αυτό ξεκάθαρα και ρητά δεν μπορεί και να λύσει το πρόβλημα. Γι' αυτό και λέω ξεκάθαρα. Ο ακροτηριασμός των γυναικείων οργάνων δεν ανήκει στην Ευρώπη ούτε και το Ισλάμ από το οποίο προέρχεται άλλωστε. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μπρούνα έχει το λόγο. 500.000 γυναίκε είναι θύματα κλειτοριδεκτομή. Ε, Αυτό ο κλητηριασμό υπάρχει στην Ευρώπη και στο έδαφο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν υπήρχε προηγουμένω στην ιστορία και τι παραδόσει των χωρών μα, ούτε στη θρησκεία και τον πολιτισμό μα. Είναι ορισμένε απομονωμένε ε, περιπτώσει του 17ου αιώνα και ήταν αυτοακροτεριασμό αυτέ οι περιπτώσει. Θα πρέπει λοιπόν να αποκλειστεί αυτή η περίπτωση από τι ομάδε των μεταναστών και επειδή δεν έχουν ε, ακόμη ενστερνιστεί τα ευρωπαϊκά ηθικά έθιμα, ε, καθώς και την παράδοσή μας. Θα πρέπει ε, ε, ο κατακλυσμός από μετανάστες που δεχόμαστε να ελεγχθεί. Υπάρχει τέτοια βάρβαρη πρακτική σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εκεί θα πρέπει να παραμείνει και όχι να εισαχθούν αυτά τα προβληματικά φαινόμενα και στην Ευρώπη, όπως με τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη προβλέπεται. Είναι εκατομμύρια γυναίκες που έχουν ε, πέσει θύματα ε, ε, στον κόσμο, να τις προστατεύσουμε στις χώρες του. Μην την εξάγουμε και εδώ ε, ω ένα πρόσθετο πρόβλημα της μετανάστευση. Ευχαριστούμε. Δεσποινής, ο κύριος Πόσπισιλ για το ΕΛΚ. Κύριε Πόσπεσου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά και υπερψήφισα το ψήφισμα αυτό, διότι η πρακτική αυτή είναι πέρα για πέρα απαράδεκτη. Πρόκειται για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήταν πολύ θετικό στη βάση αυτού του ψηφίσματο, τουλάχιστον στην Ευρώπη, να υπάρξει μια ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να επιβάλλονται και ενιαίε ποινέ εναντίον αυτών των πράξεων. Διότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο και στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Δεν μπορούμε απλά να το, κατα... να το καταδικάζουμε στα λόγια. Πρέπει με πράξεις να προσπαθήσουμε να το καταπολεμήσουμε, δηλαδή οι διοκτικές αρχές να παρακολουθούν και να διώκουν καλύτερα αυτές τις πρακτικές, να, να, τις, ε, να καταλήγουν στα δικαστήρια, γιατί αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να εξαλείψει αυτό το φαινόμενο. Σε ό,τι αφορά τις τρίτες χώρες, Θεωρώ ότι η οικονομική στήριξη και βοήθεια ε, πρέπει πάντοτε να εξαρτάται από την τήρηση των ανθρωπίνων και ιδίως των γυναικείων δικαιωμάτων. Η κυρία Τζέσικα Στέγκρουτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Τα κορίτσια ακινητοποιούνται Κατόπιν γίνεται κλειτοριδεκτομία. Στη συνέχεια γίνεται ράψιμο της ε, εγχείρησης αυτής. Αυτό αφήνει τραύματα, αφήνει πολλά προβλήματα και όταν έρθει η ώρα να γεννήσουν και σε σχέση με την περίοδό τους και σε σχέση με τη σεξουαλική ζωή τους. Πολλές φορές μολύνονται, αρρωσταίνουν, πεθαίνουν τα κορίτσια αυτά. Αυτοί οι οποίοι κάνουν τέτοια βασανιστήρια θα πρέπει να περάσουν από δίκη. Έχουν πρέσει τόσα χρόνια που έχουμε τέτοια νομοθεσία που απαγορεύει τέτοιες πράξεις στην Σουηδία. Όμως δεν έχουμε καταδικάσει κανένα και διαπιστώνεται ότι η κυβέρνηση της χώρας μας ε, δεν κάνει αρκετά και δεν τα κάνει αρκετά νωρίς. Ευχαριστώ κύριε, κυρία Πρόεδρε. Ποιο είναι το θέμα το οποίο συζητούμε σήμερα. Ποιον αφορά ο ακροτηρισμός ε, γεννητικών οργάνων. Μικρά κορίτσια 13 έως 15 ετών, χωρίς αναισθητικό, με ξηράφι, τους αφαιρείται η κλειτορίδα, τους κόβονται τα εξωτερικά χείλη του εδίου και στη συνέχεια τις ράβουν από πάνω μέχρι κάτω ώστε να παραμένει μόνο μια πολύ μικρή τρύπα. Την πρώτη νύχτα του γάμου τους ο σύζυγος παίρνει ένα μαχαίρι και κόβει τα ράματα. Αυτή την απίστευτη βαρβαρότητα την έχουν υποστεί 200 εκατομμύρια γυναίκες τον 21ο αιώνα. Και πού συμβαίνουν όλα αυτά στις Ισλαμικές χώρες. Πρέπει επιτέλους να το πούμε ανοιχτά. Διότι αυτό το φαινόμενο υπάρχει στις Ισλαμικές χώρες. Με τη μετανάστευση αυτή η απίστευτη βαρβαρότητα ήρθε και στην Ευρώπη. 600.000 θύματα, γυναίκες θύματα υπάρχουν στην Ευρώπη. Πρέπει επιτέλους να δοθεί ένα τέρμα σε αυτό το φαινόμενο. Ευχαριστούμε πολύ. Φιτζέραλτ. Σας ευχαριστώ. Εγώ ψήφισα υπέρ του ψηφίσματο. και ευτυχώς πάρα πολλοί συνάδελφοι το έκαναν αυτό. Πρόκειται για κάτι το οποίο αποτελεί βία κάθε είδους και αυτό γίνεται κατά ανηλίκων, κατά νεαρών κοριτσιών, μέχρι τα 15 αλλά και μετά 15. Έχουμε 200 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο που το έχουν ε, υποστεί. Δεν είναι κάτι που είναι μόνο στην Αφρική όπως πιστεύει ο κόσμος. Το 97% στη Γουινέα βέβαια ε, των γυναικών το πέρασε αυτό και 45% ε, κάτω από το 14% στην Ιθιοπία 65% των γυναικών, αλλά αυτό γίνεται σε χώρες σε όλο τον κόσμο, στην Ινδονησία, Μαλαισία, στην Νότια Αμερική και αλλού και στην Ευρώπη. Έχουμε 180.000 ε, κορίτσια που φοιτούν στα σχολεία μας ε, λέσχες ε, που έχουν κίνδυνο να το υποστούν αυτό. Θα πρέπει να αναλάβουμε δράση, να υπάρχει μηδενική ανοχή και χαίρομαι που υπάρχει αυτό παντού και στο νερό είδα νέους που να έχουν ταχθεί στον αγώνα κατά ε, αυτών των ακροτηριασμών. Θα πρέπει να σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο τώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα για το ECR. Η κυρία Μαργαρίτα Τελαπίσα Καριών. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Ψηφίσαμε αποχή. Είμαστε κατά του ακροτηριασμού αυτού. Αλλά δεν είναι δυνατόν αυτό να θεωρηθεί μια διακριτική μεταχείριση και να μπαίνει στο ε, ίδιο σακούλι με όλα τα άλλα προβλήματα. Το θέμα είναι ευρύτερο. Έτσι, δεν θεωρούμε ε, πρόσωπο την ε, γυναίκα. Έτσι θεωρούμε ότι δεν έχει πρωτοβουλία, δεν έχει επιθυμίες, έτσι γίνεται σκλάβα η γυναίκα. Όμως αυτό δεν το καλύπτει το κείμενο είναι κάτι πολιτιστικό, δεν είναι θέμα μόνο θρησκείας. Είναι θέμα όχι μόνο άντρα κατά γυναίκας, είναι και η γυναίκα που στρέφεται κατά γυναίκας. Και θα πρέπει να κινητοποιηθούμε ε, και όχι κατά του θεματολογίου του φεμινιστικού. Ε, θα πρέπει επομένως σε σχέση με τις δυτικές αξίες και τις χριστιανικές ε, να είναι προστατευμένη η γυναίκα. Επίγει να έχουμε ένα, μια τέτοια πηξίδα, να μην υπάρχει σύγχυση. Θα πετύχουμε μόνο αν λάβουμε υπόψη τις πραγματικές αιτίες του προβλήματος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μάριος Μπότος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα ανθρώπινα όντα δεν είναι διεκτησία κανενό. Τα παιδιά δεν είναι διεκτησία κανενό. Εδώ πρέπει να καταστήσουμε σαφέ ότι θέλουμε να θέσουμε τους δικούς μας όρους όταν μιλάμε για την προστασία των σωματών. Εκατομμύρια κορίτσια κάθε χρόνο ε, ε, απειλούνται να τους πάρουν τα δικαιώματά τους. Θα πρέπει ε, από τα 15 ε, τα κορίτσια αυτά, από τα 15 της ηλικία τους, να μην απειλούνται από γονεί, παππούδες ή κάποιον που θεωρεί στην οικογένεια ότι ωραίο είναι να περάσουν μια κλειτοριδεκτομή ή ότι πολιτιστικός αυτό είναι το δέον. Ε, πολλοί είναι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτό. Η οτι πολιτιστικό αυτο ειναι το δεον πολλοι ειναι οι κινδυνοι που σχετιζονται με αυτο η μονές ε, εξωτερική αιμορραγία, ε, θάνατο παιδιού. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να μην επιτρέψουμε τέτοια φαινομένα να εξαπλωθούν και στην Ευρώπη. Θα πρέπει ε, ο υπόλοιπο κόσμος να κοιτάξει στις, να κοιτάξει να παραμείνει το φαινόμενο στις χώρες που ο ακροτηριασμός ήδη συμβαίνει, αλλά και εκεί να καταπολεμηθεί. Εάν θέλουμε οι γυναίκες να είναι υγιεί και ισχυρά μέλη της κοινωνίας μας, αν θέλουν να γίνουν αυτές που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει και αυτές με τη σειρά τους να προστατευτούν ε, ε εκεί που πρέπει, από την αρχή δηλαδή. Ε, υπερψήφισα από το ψήφισμα και θέλετε μια καλή αρχή. Ευχαριστώ για τα λόγια σας και τώρα ο λόγια στην κυρία Βερόνικα Βρετσιόνοβα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ο ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι μια φρικαλαία ε, πράξη βίας κατά των γυναικών. Προκαλεί όχι μόνο σωματική οδύνη, αλλά και ψυχολογικά προβλήματα και προβλήματα υγείας. Είναι φρικτό στον 21ο αιώνα να ε, υπάρχουν ακόμη κράτη όπου εφαρμόζεται αυτή η πρακτική. Ε, είναι 600.000 ε, γυναίκες που πλήττονται από το φαινόμενο αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 600.000 γυναίκες που έχουν εκτηρεστεί τα γενετικά τους όργανα. 200.000 επίσης απειλούνται προσεχώς. Θέλουμε να προστατεύσουμε λοιπόν τις γυναίκες και για την ισότητα των φύλων να κοιτάξουμε να πάυσει αυτή η επονίδιστη πρακτική. Θα πρέπει να προβλέψουμε να, μην κοιτάμε μόνο τις ποσοστώσεις των γυναικών στον χώρο των πολιτικών και των επιχειρήσεων. Γι' αυτό υπερψήφισμα το ψήφισμα αυτό. αυτό. Ευχαριστούμε ο κύριος Ζαχαραντήλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε στο Ευρωκοινοβούλιο ότι είναι απαραίτητο αυτή η απάνθρωπη πρακτική να πάψει και να την καταδικάσουμε. Ε, θα ήθελα λοιπόν εδώ να επισημάνω ότι η δική μας η πολιτική ομάδα, οι συντρικοί και μεταρρυθμιστές και η δική μας ε, η κυρία Κάνκο, ε, η δική μας βουλευτής, που το 2019 ζήτησε να βραβευθεί μια ακτιβίστρια από την Κένια ε, για το κίνημα ε, εξάλληψης του ακροτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην Αφρική και στη χώρα της. Ε, εδώ λοιπόν Έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα για το θέμα αυτό και θα θέλαμε κυρία Αντιπρόεδρε να λάβετε γνώση και να να μας υποστηρίξετε εφόσον δείτε το σχέδιο αυτού του ψηφίσματος. Ευχαριστώ και με αυτό κλείνουμε τη συζήτηση για το σημείο αυτό της σημερινής διάταξης και περνάμε στο επόμενο που είναι η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Πρώτη η κυρία Πελτιέ. Η κυρία, ο κύριος Présidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού που για μένα πάει στη σωστή κατεύθυνση για την προστασία των καταναλωτών και θέλω να ζητήσω τη στήριξη του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ θα πρέπει να έχουμε συνείδηση του τι συμβαίνει με τι τεχνολογίε και την τεχνητή ευφία. Ε, δεν είναι ε, οι αλγόριθμοι σε θέση να χειριστούν ολόκληρα τις διαστάσεις της κοινωνίας μας. Ε, ο ιδιωτικός βίος, οι τραπεζικές συναλλαγές, οι αγορές. Εδώ θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο σημεία. Το κείμενο θα μπορούσε να είναι πιο φιλόδοξο στα εξή. Ως προς τη διαφάνεια που είναι μια σημαντικ... ένα σημαντικός παράγοντας για την εμπιστοσύνη των ε, συμπολιτών μας. Επίσης θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε το κείμενο προς την κατεύθυνση των λογισμικών που δεν θα πρέπει ποτέ να εξασκούν διακριτική μεταχείριση εις βάρος των πλέον ευάλωτων. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ναι στην επιστήμη, ναι στην πρόοδο, αλλά μόνο εάν συνδυαστεί με την ηθική και την ε, δεοντολογία. Ευχαριστούμε κυρία Βυσνιεύσκα. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ υπερψήφισα το ψήφισμα αυτό για να προστατευτούν οι καταναλωτές και για να προβλέπεται και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διευκολύνει τους πολίτες στην καθημερινότητά τους. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται ήδη σε διάφορους τομείς της οικονομίας και μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα. Όμως είναι σημαντικό οι εφαρμογές αυτές να είναι ασφαλείς για τους καταναλωτές και να είναι κατάλληλες για τον ε, ε, σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Και θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και για τις ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές, τις οποίες να μπορούν να ε, υιοθετήσουν. Sir, Η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σημαίνει ότι θα λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτή η απόφαση μπορεί πάντοτε να βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία, δεδομένα, ψηφιακά. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Ψηφιακό, ψηφιακή απόφαση για τη χορήγηση δανείου ή συνέντευξη για την κάλυψη μιας θέσης εργασίας. Υπάρχουν πολλά ωφέλη βεβαίως για μια τέτοια λήψη αποφάσεων. Πιο γρήγορη, και πιο εύκολη. Όμως ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Η δημιουργία προφίλ, η κατάχρηση προσωπικών δεδομένων, ο περιορισμός των καταναλωτικών επιλογών. Γι' αυτό και... Ε, Υπερψήφισα το ψήφισμα ώστε η ε, Κομισιόν να παρακολουθεί και αυτά τα ζητήματα στενά. Τόμας. Είναι πολύ σημαντικό εδώ να προσέξουμε τι θα γίνει με όλους αυτούς τους μηχανισμούς αυτοματοποιημένης λήψης των αποφάσεων. Θεωρώ ότι η τεχνολογία ήδη επηρεάζει την καθημερινή ζωή μας θετικά, αλλά θα πρέπει ξεκάθαρα να δούμε τι γίνεται, να υπάρξουν οι σωστοί αναγκαίοι μηχανισμοί για την νομοθετική ρύθμιση αυτής της διαδικασίας να προστατευτεί ο καταναλωτής. Βεβαίως και η τεχνητή νοημοσύνη κυριαρχεί παντού και είναι κάτι χρήσιμο, αλλά θα πρέπει τα παιδιά και γενικότερα οι καταναλωτές να προστατευτούν, γιατί η διαφάνεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει να μπορεί ο κόσμος να ωφεληθεί και να υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση όσον αφορά τα δεδομένα της ε, ε, τεχνητής νοημοσύνης. Περισσότερη διαφάνεια, επομένως. Επόμενος, κ. Γόλας. Η μετάβαση στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και η τεχνητή νομιμοσύνη θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίε μα και οι κατανοητέ μα λειτουργούν. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι θα προστατεύονται από αθέμητε ή διακριτικέ εμπορικέ πρακτικέ και πρέπει επίση να εξασφαλίσουμε ότι οι διαδικασίε αυτέ θα είναι διαφανεί και δεν θα συμπεριλαμβάνουν δημιουργία προφίλ. Από αυτή την άποψη, η παρακολούθηση τη αυτοποιημένη λήψη αποφάσεων θα πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητου τρίτου φορεί. Θα πρέπει να μπορεί κανεί να υποβάλει ένσταση ε, σε περίπτωση λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων. Θα πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να εξασφαλίσει ότι τα πλαίσια που θεσπίζονται είναι κατάλληλα για τον, για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Οι αρχέ θα πρέπει να είναι, αρκε... Ε, να είναι επαρκώ Δεν μπορούμε να αφήσουμε την, ε, τις αποφάσεις αυτές σε μια χούφτα εταιρείε που θα ελέγχουν τον κλάδο αυτό. Θα πρέπει πάντοτε να τηρούνται οι αρχέ του Γενικού Κανονισμού Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κλούιν εκ μέρου του ΕΛΚ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Η τεχνητή νοημοσύνη δίνει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται κανεί πολύ περισσότερα δεδομένα από ό,τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι σε ένα κλάσμα αυτού του χρόνου. Είναι μια πρακτική η οποία χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στο νομικό σύστημα, στην ε, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Οι αλγόριθμοι πολλές φορές όμως μπορούν να έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά την πρόσβαση ανθρώπων σε ε, νομικές υπηρεσίες, υγειονομικές υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Εγώ λοιπόν με χαρά υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα που καλεί την Κομισιόν να εξετάσει αν χρειάζονται περαιτέρω βήματα για να προστατευτούν τα δικαιώματα των καταναλωτών στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, να προστατεύονται από αυθαίρετες και διακριτικές ε, συμπεριφορές ή αποφάσεις, να ενισχυθεί η διαφάνεια και να εξασφαλιστεί ότι μόνο ε, υψηλή ε, ποιότητας και όχι μεροληπτικά σύνολα δεδομένων θα χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Σε τελική ανάλυση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, εξασφαλίσει ότι οι όροι και οι κανόνες της είναι κατάλληλοι για, το, για την ψηφιακή εποχή. Ευχαριστώ. Και τώρα μιλάμε, θα μιλήσουμε για την ε, νέα σχέση με, την, ε, με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και, του, και της Βόρειας Ιρλανδίας. Ο συνάδελφος Σκέλεχερ έχει το, πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω εξ αρχής ε, ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, ιδίως στο πλαίσιο της Ιρλανδίας. Οι πολίτες στην Βόρεια Ιρλανδία ενδιαφέρονται πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Όσον αφορά δηλαδή την θέσπιση τη σύναψη μια εμπορική συμφωνία Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε πάντοτε στο επίκεντρο τη προσοχή μα του Ιρλανδού πολίτε. Υπάρχουν εκατοντάδε χιλιάδε Ιρλανδοί πολίτε που είναι πολίτε βεβαίω τη Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίοι αυτή τη στιγμή ζουν στην Βόρεια Ιρλανδία εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιστεύω ότι όταν συζητάμε αυτά τα θέματα και δεν ζητώ καθόλου συγγνώμη για το γεγονό ότι διαρκώς ε, επιμένω στις ανησυχίε των ε, Ιρλανδών ε, που ζουν στην Βόρεια Ιρλανδία. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί η Συμφωνία τη μεγάλη παρασκευή, σε οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία στο μέλλον. Η αναγνώριση προσόντων, για παράδειγμα, είναι ένα από τα σημεία οποία θα πρέπει να, στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι άνθρωποι και από τις δύο πλευρές των συνόρων να μπορούν να εργάζονται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων στο νησί της Ιρλανδίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαριανή έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι Βρετανοί συναδελφοί έφυγαν. Θα πρέπει να μην ξεχάσουμε τον κύριο Φάραζο διότι ήταν το ε, σύμβολο ε, του πατριώτη της εθνικής ταυτότητας κόντρα σε όλους ήθελαν να σβήσουν όλα αυτά ε, τώρα θα πρέπει να δούμε τι, τι δομή θα έχουν τα θεσμικά όργανα και θα πρέπει ε, κόντρα σε αυτό το ψήφισμα να, να μην φυγεί η εθνική κυριαρχία για την ε, Βρετανία. θεωρούσαν ότι δεν υπήρχε ισορροπία μεταξύ των εθνών, δεν υπήρχε ισορροπία μεταξύ των πλειονεκτημάτων, των στόχων, των μέσων ε, που χρησιμοποιούνται μέσα σε αυτή την κατάσταση ε, οπότε αυτό ήταν ένα δίδαγμα που μας έδωσαν κάποιες προσωπικότητες της ε, Βρετανίας θα πρέπει να τους σεβαστούμε και γι' αυτό το λόγο εγώ απέσχων από την ψήφιση. Και τώρα για το ΕΛΚΑ. Ε, κυρία Φιτζέρλ. Σας ευχαριστώ. Ψήφισα ε, ε, αυτό το κείμενο το οποίο καθορίζει την μέλουσα σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με το Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά θα πρέπει να κλειστεί αυτή η εμπορική συμφωνία. Θα πρέπει να έχουμε όσο γίνεται πιο σωστή θέση και να κατοχυρωθεί και uh, να αυτό να γίνει με σεβασμό θα, θα πρέπει να ακούμε αυτά τα διαφορούμενα που ακούμε από το Ευρωπαϊκό, από το Ηνωμένο Βασίλειο και να δούμε τι θα έχει με τη Βόρεια Ιρλανδία. Οπότε είναι θετικό αυτό που λέει το κείμενο, ότι θα πρέπει η μέλουσα σχέση να βασίζεται στην ισονομία όσον αφορά τις οικονομικές εταιρικές σχέσεις και άρα έτσι να εξασφαλιστεί μια σχέση που θα τους βρίσκει όλους κερδισμένους. Έχουμε πολύ εμπόριο με τη χώρα, αλλά επίσης θα πρέπει να προστατευτεί και η ειρήνη στην Βόρεια Ιρλανδία. Ε, με, να μην ε, τεθεί ένα αμφιβόλο η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, ότι ρυθμιστεί δεν θα πρέπει να αναιρεί συμφωνήσαμε προηγουμένως ε, και στη συμφωνία της αποχώρησης. Αυτό θα πρέπει να μας προσβεί στους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα θα έχει τον λόγο η κυρία Βυσνιεύσκα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά το Brexit, οι σχέσεις ε, Βρετανίας και Ένωσης θα πρέπει κάπως να ρυθμιστούν και ακριβώς ε, με αυτό το ψήφισμα Έχουμε τις ε, συστάσεις προς την Κομισιόν για τις διαπραγματεύσεις. Εδώ έχουμε μια σειρά από πολιτικές, ε, τρεις βασικούς ε, άξονες, οικονομικά, τομεακά, θεματική συνεργασία και καλύπτουμε και την συνεργασία σε άμυνα και εξωτερική πολιτική. Εννοείται ότι μια χώρα που δεν είναι κράτος μέλος δεν μπορεί να έχει τα ίδια δικαιώματα, προνόμια με τα κράτη-μέλη. Αλλά να θυμόμαστε ότι η μέλουσα σχέση μας θα πρέπει να είναι ε, κάτι που να βασίζεται σε πνεύμα συνεργασίας. Έχουμε δεσμούς ιστορικούς και οικονομικούς με την χώρα. Επομένως, είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών να έχουμε τις καλύτερε δυνατές σχέσεις. Γι' αυτό και ψήφισα υπέρ η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Η κυρία Σόιντροβα για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρόλο που δεν συμφωνώ και δεν, επιθυμώ την, δεν επιθυμούσα την αποχώρηση της του Ηνωμένου Βασιλείου, της Μεγάλης Βρετανίας ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει διευθέτηση της εταιρικής μας σχέσης και της μελλοντική σχέσης μεταξύ των κρατών μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό λοιπόν το Ευρωκοινοβούλιο ε, μέσω των ε, πολιτών ευρωπαϊκών δεσμών των ευρωπαϊκών κρατών προς το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει ενωμένο. Και συμφωνούμε πιστεύω όλοι ότι η κοινή μας δουλειά θα πρέπει να καταλήξει σε μια αίσια έκβαση. Εδώ ε, λαμβάνουμε γνώση του γεγονότος ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει μια σχέση τρίτου κράτους και ελεύθερων συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει η φραγμή είναι ενός το δυνατόν ε, λιγότερη. Θα πρέπει η κυκλοφορία των αγαθών και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά να σέβονται όλα τα κριτήρια ποιότητας, ε, τις ενδείξεις, τη χρήση φυτορμάκων για τα τρόφιμα και το καθεξής, να τα λαμβάνουν υπόψη και να γίνονται σεβαστά. Θα πρέπει να προστατευτούν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι Ευρωπαίοι πολίτες επίσης. Ευχαριστούμε και τώρα ο κύριος Πόσπιφιλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ ε, και εγώ ε, υποστήριξα αυτή τη διαπραγματευτική εντολή γιατί θεωρώ σημαντικό τουλάχιστον δύο πράγματα να γίνουν οπωσδήποτε. Πρώτα απ' όλα τα δικαιώματα των ε, πολιτών μας στην Μεγάλη Βρετανία και αντιστρόφως να προστατευθούν. Επίσης θεωρούμε ότι η συμφωνία αυτή ε, πρέπει να ε, ε, καλύψει τα δικαιώματα όλων. 30.000 Τσέχοι ζουν ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει εδώ λοιπόν να υποστηριχθούν. Και η συμφωνία για, ελεύθερες, για για με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σημαντικό για να προστατευτούν οι εξαγωγέ και από τι δύο πλευρέ και να γίνονται σεβαστέ όλε οι προποθέσει τη εσωτερική αγορά. και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσει προβλήματα το Brexit. Είναι πολλέ τσεχικές εταιρείε που εξάγουν προ το Ηνωμένο Βασίλειο και θα πρέπει όλα να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε οι βασικές προϋποθέσεις να γίνουν σεβαστές. Ο κύριος Μπομπάρ. Κύριε Πόλτσακ, σας ξέχασα. Με συγχωρείτε. Ευχαριστώ, το Brexit δυστυχώς για μένα ήταν πολύ ατυχές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Μεγάλη Βρετανία βέβαια το έτσι ως επιτυχία. Εδώ λοιπόν υπερψήφισα αυτή τη συμφωνία για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι ο κίνδυνος ενός σκληρού Brexit ακόμα δεν έχει αποφευθεί πλήρως. Δυστυχώς ο Βρετανός Πρωθυπουργό έχει εξηγήσει ότι οι διαπραγματεύσεις μετά το Brexit θα πάνε στην πορεία που θέλει εκείνος. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε με κάθε τίμημα να παραμείνουμε ενωμένοι και ενιαίοι στην ε, στάση μας. Θα πρέπει να φροντίσουμε να προστατευτούν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών αλλά και τη ε, δημοκρατία τη Ιρλανδία, τη Βόρεια Ιρλανδία. Η κυκλοφορία των ε, αγαθών και των υπηρεσιών. Θα πρέπει όλα να τα παρακολουθήσουμε προσεκτικά. Και υπάρχει και ένα ε, ραντεβού στο τέλο τη χρονιά για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει και τα περιφερειακά κοινοβούλια να έχουν ε, συμμετοχή και να προστατευτούν και οι δικές τους επιθυμίες. Ευχαριστούμε και τώρα ο κύριος Μπομπάχα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτή η εντολή πρόκειται να οδηγήσει στην πιο μεγάλη εμπορική συμφωνία που έχει ποτέ συνάψει η Ευρώπη. Και όπως πάντα ε, πρόκειτο για ε, καλή πίστη και για κάποιους ευσεβείς πόθους. Αλλά δεν είμαστε χαζοί γιατί μπροστά από αυτή την ε, βιτρίνα υπάρχει καθήλωση στον φιλελευθερισμό που μας καταστρέφει το περιβάλλον, καταστρέφει τον κόσμο, τα ιδιωτικά δικαστήρια, προσήλωση σε ποσοστώσεις ε, μηχανισμοί της αγοράς για να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση. Επομένως πρόκειται για ε, προσήλωση στο ΝΑΤΟ και στην στρατικοποίηση. Συνάδελφοι, ε, μόλις έφυγαν οι Βρετανοί και όλα συνεχίζονται όπως πριν. Μα τότε τι θέλετε ούτω άστε τελικά να μάθει το μάθημά του το κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ λέει η πρόεδρος και τώρα έχουμε τον κύριο Κιουτσούκ. Σας ευχαριστώ. Ε, κυρία Πρόεδρε. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα και δεν ακούγεται ο μιλητής. Πρόκειται για κάποια κοινή θέση που θέλουμε να υιοθετήσουμε συνεχίζεται το πρόβλημα. Thank you very much. We just realized it. Thank you very much. Okay. Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ του κειμένου. Χρειάζεται μια σφαιρική συμφωνία με την Βρετανία. Πιστεύουμε ότι πρέπει να μπει ψηλά ο πύχης για την εταιρική σχέση και έχουμε διάφορα επιμέρους θέματα. Θέλουμε να είναι μια συμφωνία που να μην περιέχει δασμούς αλλά να μην οδηγήσει και σε dumping. Δεν θέλουμε πρότυπα συμφωνίας με Καναδά και Αυστραλία όπως λέει ο Τζόνσον. Θα πρέπει να ισχύσουν τα όσα ορίζει ο ΠΟΕ. Ό,τι συμφωνία και να γίνει με την Βρετανία θα παραμείνει τρίτη χώρα. Άρα θα πρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία μας πάνω από όλα. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ και τώρα ο κύριος Τόματς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου μιλάμε για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τώρα πρέπει να ε, χτίσουμε μαζί τους μια ειδική σχέση. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε τουλάχιστον δύο πτυχές. Πρώτον, υπάρχουν πολλοί Βρετανοί που οδέποτε θέλησαν ε, το Ηνωμένο Βασίλειο να καταλήψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κατά δεύτερον, υπάρχουν 3,5 ε, εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα. Αυτό αυτοί δεν θα πρέπει να πληγούν από τις λαϊκιστικές πολιτικές που ήθελε να, που έφεραν το Ηνωμένο Βασίλειο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως κάποια μέρα το Ηνωμένο Βασίλειο να ξανάρθει στους κόλπους της Ένωσης. Με συγχωρείτε ε, που σας διακόπτω, αλλά ο κύριος ε, Μπλέτς, ε, ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Έχουμε δει ποιε θα είναι οι επιπτώσει ε, του Brexit αν υπάρξουν ομαλέ διαπραγματεύσει. Το έχουμε σκεφτεί. Αλλά τι θα γίνει αν υπάρξει ένα σκληρό Brexit. Θα πρέπει να το αποφύγουμε και το Κοινοβούλιο να παίξει εδώ ένα ενεργό ρόλο. Θα πρέπει το θεσμικό μα όργανο που είναι απευθεία εκλεγμένο από του πολίτε να κάνει ό,τι μπορεί. Και εμεί να βεβαιωθούμε τα δικαιώματα των πολιτών γίνονται σεβαστά. Η νέα εντολή είναι καλή. Είναι κάτι το θετικό γιατί αναφέρει τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την ε, υπάρχουσα σχέση μας και εξηγεί ότι η νέα σχέση θα είναι διαφορετική από τη σχέση ενός κράτους μέλους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή Απασχόλησης έχει τοποθετηθεί σχετικά και η άποψή της έχει ληφθεί υπόψη. Θα πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινε γραμμέ μα όταν θα πρέπει να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μα. Ευχαριστούμε και τώρα από του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ, ο κύριο Ρόντσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κυρίες και κύριοι, εδώ μιλούμε για μια κατάσταση άνευ προηγουμένου και άγνωστη ως τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον πιο αδύναμη και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Ε, και ειλικρινώς. Τώρα όμως ξεκινούμε συζήτηση για τη μελλοντική ε, σχέση και συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Πραγματικά εύχομαι ο κύριος Μπαρνιέ να τα καταφέρει και η συμφωνία αυτή να είναι η βέλτιστη δυνατή. Ωστόσο, όλοι ε, θέλουμε και επιθυμούμε να υπάρξουν ε, καλές, ομαλές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι σημαντικό είναι σημαντικό να κατασβεστεί αυτή η πυρκαγιά και να λάβουμε μέτρα ε, και για το μέλλον. Θα πρέπει να φροντίσουμε την ασφάλειά μας στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο και να μην το ξεχνάμε. Χρειαζόμαστε ένα κόσμο ασφάλειας και μια ασφαλή Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Και τώρα για το ΕΛΚ η κυρία Κλούν. Ε, Ευχαριστώ αυτή η μέλουσα εμπορική συμφωνία όποτε και εάν ολοκληρωθεί θα πρέπει να περάσει από το Κοινοβούλιο οπότε είναι θετικό αυτό το ψήφισμα ε, είπα ναι σε αυτό έχουμε τις προτεραιότητές μας ό,τι θέλουμε να καλύψει η συμφωνία ιδίω δε τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και τη ρύθμιση που θέλουμε για το καθεστώς που θέλουμε να προστατεύσουμε εμπόριο ε, διέλευση με το Ηνωμένο Βασίλειο οπότε αυτά θα διέπουν την διαπραγματευτική εντολή και χρειάζεται και για τις δύο πλευρές μια συμφωνία από την οποία να είναι όλοι κερδισμένοι, να μην βγουν χαμένες οι εταιρείε μας άρα θα πρέπει να προστατεύσουμε τους καταναλωτάς επίσης και αυτό θα γίνει μα είμαστε η έκτη πρόκειται για στην Βρετανία η έκτη μεγαλύτερη δημορική δύναμη και πρώην ε, μέλος της Ένωσης ή πρόεδρος Σικόρσκι, ε, παρακαλώ για το ΕΛΚ ένα λεπτό ψήφισε. Η Πρόεδρε, ψήφισα την ε, συμφωνία γιατί προστατεύει επαρκώς τα συμφέροντά μας αλλά δεδομένης της συμφωνίας και των κόκκινων γραμμών της Βρετανικής κυβέρνησης που δεν θέλει τελωνιακή ένωση ε, δεν θέλει δικαιοδοσία του ΔΕΚ και δεν θέλει ελεύθερη μετακίνηση ε, έχουμε μια ελάχιστη συμφωνία για τα αγαθά και η πυραμίδα του ψέματος των ευρωφοβικών στην Βρετανία έχει αρχίσει να καταραίει. Η Βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι θα υπάρχουν τελωνιακοί και άλλοι έλεγχοι στα σύνορα. Άρα, στο όνομα του ελευθέρου εμπορίου, η Βρετανία θα εγείρει εμπόδια στον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της. Οποία καταστροφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τελειώσουμε τον κύριο Σόνκελ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ σημαντικό αυτό ψήφισμα είναι ένα βασικό βήμα για το ξεκίνημα των διαπραγματεύσεων. Είναι πολύ θετικό το ότι εδώ πέρα αντικατοπτρίζεται μια μεγάλη φιλοδοξία για μια ευρεία συνεργασία με το Ερμένο Βασίλειο. Επίσης, θα πρέπει να συνεχίσει η αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας αυτής σε αποχώρησης μαζί με τις διαπραγματεύσεις. Επίσης ε, δίνουμε βάρος ε, στο να προστατεύσουμε την Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και τη κοινού χώρου ταξιδίων, κάτι τα οποία ε, είναι βασικές προτεραιότητες για την Ιρλανδία και για τους 27. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την στήριξή τους και ελπίζω να έχουμε ε, ειλικρινή συνεργασία από το Ηνωμένο Βασίλειο για να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώθηκε αυτός ο γύρος. Και περνάμε στην έκθεση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μικ Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ιρλανδική Κεντρική τράπεζα ακόμα ξεπληρώνει τα 31 δισεκατομμύρια ευρώ από τα ομόλογα από την καταστροφή του 2008. Οι τράπεζες ε, τελικά έκλεισαν, αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιμένει να εξοφλήσει τα 31 δισεκατομμύρια η Κεντρική Τράπεζα. Υποφέραμε μία δεκαετία λιτότητας, ε, στην οποία πρωτοστάτησε η κυρία Λαγκάρντ. και βεβαίως ε, και ο κύριος Ντράγκη το εκμεταλλεύτηκε για το δημοσιονομικό του σύμφωνο το οποίο θεσμοποίησε την λιτότητα. Πρόκειτο λοιπόν για ένα νέο όνειρο, τον απόλυτο διαχωρισμό της δημοκρατικής διαδικασίας από την ε, οικονομική πολιτική. Όπως είπε και ο Γερμανός ε, Υπουργός Οικονομικών του 2015, οι εκλογές δεν αλλάζουν τίποτα. Υπάρχουν κανόνες. Δεν θυμάμαι λοιπόν καμία έκθεση τη ε, ΕΚΤ να τα αναφέρει αυτά και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε ποτέ. Βεβαίως είμαστε κατά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Βάιμερς για το ΙΣΙΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η Σουηδία πρέπει να πει όχι στο ευρώ. Στην έκθεση μάλιστα α, μας λέει η Κεντρική Τράπεζα ότι είναι υποχρεωτικό να υιοθετήσουμε το κοινό νόμισμα. Κοιτάξτε, εμείς κάναμε δημοψήφισμα και η πλειοψηφία ήταν κατά. Τώρα, γνωρίζουμε πως υπάρχουν πέντε χώρες που δεν έχουν το ευρώ. Γνωρίζουμε πως ε, το χρήμα διασχίζει τα σύνορα και είναι δύσκολο βεβαίω όταν υπάρχουν διαφορετικά νομίσματα. Θέλουμε την Σουηδική κορώνα. Πόσο δύσκολο είναι να το καταλάβετε. Λέτε ότι είστε δημοκράτε, αλλά δεν έχετε κανένα σεβασμό στην βούληση του λαού. Έχουμε μια δύναμη κυβέρνηση η οποία δεν διαπραγματεύτηκε opt-out από το ευρώ. Δεν το θέλουμε το ευρώ. Και θα φροντίσουμε να πάρουμε opt-out. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ομπρή. Εδώ και μερικού μήνε όλοι χειροκροτούσαν το διορισμό μια γυναίκα επικεφαλή Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ε, Όμω, ε, αλλά είναι, το δάσο που κρύβει το, το δέντρο που κρύβει το δάσο. Ο σεξισμό εξακολουθεί να υπάρχει. Φέρα εδώ μερικέ φωτογραφίε αυτών που αποφασίζουν σήμερα για την οικονομική και νομισματική διακυβέρνηση τη Ευρώπη το διευθυντικό ε, όργανο της ε, ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μόνο δύο γυναίκες. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επίσης το ίδιο. Ελάχιστες είναι οι γυναίκες και αυτές γιατί δεν υπάρχουν επαρκώς ε, ικανές γυναίκες για να λάβουν αυτές τις θέσεις. Θα πρέπει να πάρουμε μέτρα ε, έτσι ώστε να γίνει υποχρεωτική η ε, εξίσωση των γυναικών με τους ε, άντρες. Εμείς δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ντάλη από την ΚΟΕ. Με χαρά είδα την κυρία Δαγκάρντ εδώ αλλά με απογοήτευσε το γεγονό ότι δεν κατάφερα να μιλήσω, να πάρω το λόγο. Στην Ιρλανδία είναι πολύ γνωστή για το ρόλο της στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τα άγρια μετραλιτότητας που επέβαλε. Το αποτέλεσμα ήταν μια χαμένη δεκαετία. Το bailout ήταν ε, 64 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά το ανθρώπινο, η ανθρώπινη ζημιά είναι πολύ μεγάλη και πληρώνεται ακόμα. Ε, παιδιά που δεν τρέφονται σωστά, ε, άντρες και γυναίκες που χάνουν τη ζωή τους στο νοσοκομείο. Ε, την περασμένη, το περασμένο Σαββατοκύριακο όμως οι Ιρλανδοί πολίτες έδωσαν την απάντηση ότι που η Φίνα Φιόλ και η Φίνα Γκέλ που ήταν τα δύο κυβερνητικά κόμματα που ήταν υπεύθυνα για αυτή την κρίση πήραν το μάθημά τους εκλογές. Ο νεοφιλελευθερισμός βρίσκεται στο, στην καρδιά τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δεν θα τον δεχτούν οι πολίτε μα. Ευχαριστώ. Σίλβια Μόντικ. Πρόεδρε, το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα της ζώνης του ευρώ είναι το σύμφωνο σταθερότητας. Ε, το οποίο καθιστά δυνατές ε, τις ε, προκυκλικές πολιτικές και καθιστά αδύνατες τις επενδύσεις στο κλίμα και στην ουδέτερη πλευρά άνθρακα οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όμως έχει ως τμήμα της εντολής της να συμμετάσχει και να συνεισφέρει στην ε, ε, καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Η κρίση που μας περιμένει εξαιτίας αυτού, εξαιτίας της ε, μείωσης της του άνθρακα είναι μεγάλο πρόβλημα για το μέλλον. θα έπρεπε τώρα να αφιερώσουμε πολύ μεγάλα ποσά στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Ένα από τα σημεία τα οποία κρεμούν είναι τα πράσινα ομόλογα τα οποία θα πρέπει να μπορεί να αγοράσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Δυστυχώ δεν καταφέραμε να το κάνουμε αποδεκτό.